στο τέλος της συζητήσεως και μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης δηλώσει Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της καταστάσεως στην Ονδούρα. Πρώτος αγορητής εκ μέλους του Συμβουλίου είναι ο υπουργό ο κύριος Μπίλτ. Ευχαριστώ. Ο κόσμος είναι μεγάλος κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να επικεντρωθώ κάπως στην υπόθεση της Ονδούρας. Έχουμε μια σειρά εξελίξεων εκεί, όχι μόνο στις Ονδούρας, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σχετικά σύντομος. Στην... Ξεκίνησε η κρίση τον προηγούμενο μήνα και η Προεδρία καταδίκασε το στρατιωτικό κίνημα κατά του Προέδρου Μαρία ε, αυτή η δράση παρέμβαινε το συνταγματική τάξη της Ονδούρας. Ζητήσαμε την αποκατάσταση λοιπόν του κράτους δικαίου, συνταγματικού καθεστώτος πλήρως και ζητήσαμε από όλα τα κόμματα και τους θεσμούς να αποφύγουν τη βία, τη συζήτηση για βία και να προσπαθήσουν να βρουν μια γρήγορη και ειρηνική λύση. Νομίζω ότι λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο όπως αναμένουμε όταν εμφανίζονται προβλήματα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης ε, ε, περιμένουμε σε αυτές τις περιπτώσεις η Ένωση να ηγηθεί των προσπαθειών και εμείς τώρα ελπίζουμε ότι ο υπόλοιπο κόσμος θα υποστηρίξει την προσπάθειά μας ώστε να εξευρεθεί μια λύση διαλόγου και συμβιβασμού για την επίλυση των προβλημάτων που ε, εμφανίζονται. Κανένας από τους πρέσβεις μας που βρίσκονται επί τόπου ε, ε, μάλλον κανένας από τους πρέσβεις μας δεν είναι παρόν στις, επιτόπου αυτή την εποχή και δεν έχουμε διπλωματικές επαφές. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Κωνσταντίνα και για το βραβείο Νόμπελ που προσπαθεί να συμφιλιώσει τις ε, προσπάθειες εκεί. Είναι δύσκολο όμως το εγχείρημα, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξουν ε, νέες ε, συναντήσεις αυτό το Σάββατο κάτω από την Προεδρία του Προέδρου Αρίας. Τον παροτρύνουμε λοιπόν να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειές του και παροτρύνουμε και τις δύο πλευρές να προσπαθήσουν να συμβιβαστούν σεβόμενοι κάθε άρθρο του συντάγματος των Ονδούρας. Θα ήθελα ακόμη να υπογραμμίσω την σπουδαιότητα την οποία αποδίδουμε ε, πέραν της σημερινής κρίσης την οργάνωση διαφανών προεδρικών εκλογών στις Ονδούρες το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι ο κραγωνιαίος λίθος της δημοκρατικής κυβέρνησης, κάθε δημοκρατικής κυβέρνησης. Σε όλη την Αμερική δεν εξαιρείται καμία χώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο εκπρόσωπο της Κομισιόν, η κυρία Κατερίνα Άστον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι τα μέλη του Κοινοβουλίου και με χαρά θα συμβάλλω σύντομα σε αυτή τη συζήτηση εκ μέρους της ε, συναδέλφου Βάλνερ ε, εξετάζοντας την πολιτική κρίση της Ονδούρας. Πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια μάλλον, έχουμε συνταγματική ρήξη στη Λατινική Αμερική. Οι κρίση στις Ονδούρες μας δείχνουν πόσο εύθραυστο είναι το κράτος δικαίου και το συνταγματικό πλαίσιο για την επίλυση συγκρούσεων στις λατινοαμερικανικές χώρες. Δηλαδή αυτές οι χώρες μπαίνουν, βυθίζονται σε κρίσει, ιδιαίτερα τώρα που αντιμετωπίζουν πόλωση, έντονη πόλωση πολιτική. Η Κομισιόν αντέδρασε σωστά. Άμεσα διατυπώσαμε την ανησυχία μας, τονίσαμε πόσο απαραίτητος είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των συνταγματικών θεσμών και επιμείναμε προς όλα τα κόμματα να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά, σεβόμενοι το νομικό πλαίσιο της χώρας τους, ξεκινώντας ένα διάλογο για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη χώρα. Καταγγείλαμε τις βίες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα καθώς έχουν οδηγήσει στην απώλεια ανθρώπινης ζωής, και ζητήσαμε από όλες τις πλευρές να είναι μετριοπαθείς. Η Κομισιόν δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κατατείνει σε μια ειρηνική λύση της κρίσης για την αποκατάσταση του συνταγματικού πλαισίου. Υποστηρίξαμε την πρωτοβουλία της ε, οργάνωσης των Αμερικανικών κρατών και του κυρίου Σούλτσα, του Προέδρου. Δυστυχώς η πρωτοβουλία αυτή δεν απέδωσε. Καλωσορίσαμε και τις ε, διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Προέδρου της Κωνσταντίνα και φαντάζομαι ότι μπορεί να οδηγήσουν σε ειρηνική λύση. Μετά τα γεγονότα στις Οντούρες και αφού ήρθαμε σε επαφή με τις κέντροαμερικανικές κυβερνήσεις αποφασίσαμε να σταματήσουμε την συνέχιση ε, των διαπραγματεύσεων με την Κεντρική Αμερική. Επρόκειτο να γίνουν 5 με 10 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις αυτές όμως βεβαίως μπορούν να ξαναρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν. Όπως είπε και η Προεδρία σε σχέση με τη σοβαρότητα της υπόθεσης ε, έχουμε ανακαλέσει τους πρέσβεις σε στενή συνεργασία με την Προεδρία και τα κράτη-μέλη συνεχίσαμε να διερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε καλύτερα να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτής της κρίσης. Προς το παρόν η αναστολή της συνεργασίας δεν έχει αποφασιστεί αλλά η καταβολή δημοσιονομικών υποχρεώσεων έχει ε, ανασταλεί. Τα γεγονότα στις οντούρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αποτελέσουν με συγχωρείτε, ε, μία υπαναχώρηση, ένα βήμα προς τα πίσω και να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Γι' αυτό παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και υποστηρίζουμε κάθε επιπροσπάθεια για μια ειρηνική λύση. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για οποιασδήποτε εξελίξεις. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Θα ακούσουμε πρώτα τους ομιλητές εξ ονόματος των διαφόρων πολιτικών ομάδων και πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Αλαφράκα εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάνου Μιλιτάρη τον έβαλαν από το σπίτι του, τον πρόεδρο, τον εκλεγμένο. Και τον έβαλαν σε ένα αεροπλάνο για να τον ε, μεταγάγουν σε ξένο κράτος. Αυτό θα πρέπει ε, απερίφραστα να καταδικαστεί από δημοκρατική πλευρά. Και με βάση όλα αυτά κύριε Πρόεδρε πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαν πολλοί αναλυτές ε, εξέχοντε, όπω ο συγγραφέα Μάριος, ε, Μάριο Βάργας Λιώσα. Ο πρόεδρος Πελάγια έχει συγκεντρώσει το πρόσωπό του ομοφωνία των διαφόρων πολιτικών ε, κομμάτων και του συνταγματικού δικαστηρίου και βλέπουμε όμως τα καθεστώτα αυτά συστηματική ε, περιστολή των ελευθεριών, της δημοκρατίας, όπως είπε και το Κοινοβούλιο στην τελευταία του έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Τώρα θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Το είπε και ο Προεδρεύων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτρέψει και να διευκολύνει επάνωδο στη δημοκρατική ομαλότητα και επιπλέον ο άνθρωπος αυτός βοήθησε και τον Όσκαρ Άρια στην Κωνσταντίνα για να εξομαλωθεί η κατάσταση στην περιοχή. Θα πρέπει στη χώρα ε, να θέσουμε να δώσουμε όση βοήθεια μπορούμε με παρατήρηση των εκλογών και με βοήθεια για τη διεξαγωγή των εκλογών σε τεχνικό επίπεδο και εμπειρογνωμών. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να ενισχύουμε την πολιτική και γενικότερη συνεργασία μας με τη μόνη μη δημοκρατική χώρα της περιοχής και αφήνουμε τους υπολείπους στη μοίρα του. Και κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως είπε ο κύριος Μπίλτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ενεργό ε, παρουσία στην περιοχή. Αυτό το καιρό ε, έχει διαπραγματεύσει τη συμφωνία σύνδεσης που ολοκληρώνεται σε λίγο και δεν μπορούμε να αφήσουμε μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά και να την πληρώσουν κάποιοι αθώοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράκα. Εξ ονόματος Σοσιαλιστικής Ομάδας για 1,5 λεπτό έχει ο κύριος Γενιές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην ομόφωνη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας προσθέτουμε και εμείς τη φωνή μας, όχι απλώς επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα, όπως είπε και ο Προεδρεύων και η Επίτροπος, για την κατάσταση αυτή καθ' αυτή, δηλαδή ότι ε, έχει καταληθεί η δημοκρατική συνταγματική τάξη, αλλά είναι και σημαντικότατο προηγούμενο σε μια περιοχή που με πολλή δουλειά και με πολλή προσπάθεια κατάφερε να ξαναφέρει τη δημοκρατία σε όλη την Ήπειρο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε εμεί να διαφορήσουμε. Καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ανακαλέσουν του πρέσβει και να ακυρώσουν κάθε είδου συνεργασία, να ανασταλούν και οι διαπραγματεύσει με την περιοχή. Τώρα όμω θα πρέπει να υποστηρίξουμε και συμφωνώ με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία έξοδο μέσα από διάλογο. Ο Σκαράριας, ε, ε, που έχει βραβευτεί με τον Ρόμπερ και είναι και σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο στην Κωνσταντίνα, σε αυτή την ε, κατάσταση. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να αναλύουμε τα σφάλματα πραγματικά υποτιθέμενα που έχει ε, κάνει ενδεχομένω και ο πρόεδρος Σελάγια. που είχε έξι μήνες για να ολοκληρώσει τη θητεία του. Τώρα είναι η στιγμή της ανάλυσης του σοβαρότατου αυτού πλήγματος ε, στην ένωμη τάξη ε, και τη συνταγματική από πλευράς του στρατού Βέβαια υποστηρίζεται και από το Κογκρέσο και από ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά αυτά είναι τελείως παράνομα και ε, εξωφρενικά. Θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του Προέδρου Σελάγια, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψει ο εκλεγμένος ε, συνταγματικός πρόεδρος στη χώρα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2010. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, το λόγο έχει η κυρία Ισάσκουν Μπιλμπάου την οποία καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο ημικύκλιο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, ε, χάρη σε εσάς. Ε, καλησπέρα σας και ε, σε όλους ε, θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Μιλώ βασικά. Είναι μια γλώσσα μειονοτική η οποία δεν είναι επίσημη ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω και στο μέλλον να μπορέσει να γίνει όπως και άλλες γλώσσες και να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε την μητρική μου γλώσσα, τη γλώσσα της χώρας των Βάσκων. Θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα μου και εγώ καταδικάζουμε το πραξικόπημα αυτό, γιατί θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό έγινε στην Ονδούρα. Ορισμένοι μπορεί να το θεωρούν αυτό σφάλμα και δεν θα το αναλύσουμε Ίσως δεν δόθηκε στο λαό η ευκαιρία να κάνει τη φωνή του να ακουστεί, αλλά τώρα θα πρέπει να επανέλθει η συνταγματική τάξη και η θεσμική τάξη μετά από αυτό το πλήγμα που δέχτηκε και να επιστρέψει ο πρόεδρος της Ονδούρας στη χώρα του. Εξελέγει νόμιμα από όλου τους πολίτες. Επίσης, συμμερίζομαι την ανησυχία ορισμένων υπουργών και διπλωματικών αντιπροσωπιών, όπως ακούσαμε έχουν ανακληθεί πολλοί πρέσβεις και βεβαίως και η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει όλες τις δράσεις, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, των Αμερικανικών κρατών για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση στη ε, σύγκρουση αυτή. Η ομάδα μου επιθυμεί να εκφράσει και αυτή την επιθυμία της. Δηλαδή ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την δημοκρατική τάξη στην Ονδούρα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τελικά ο πολιτικός διάλογος να είναι το μόνο μέσο που θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα να στηρίξω και τον κύριο Όσκαρ Αρίας, που έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, στις προσπάθειές του και ελπίζουμε το Νοέμβριο του 2009 να γίνουν εκλογές σε πλήρη διαφάνεια και σεβασμό της δημοκρατίας, του δημοκρατικού συστήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελπίζω να μπορέσουν να συνεχιστούν και οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την γενναιοδορία σας. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ρωμέβα η Ρουέδα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ επ' ευκαιρία να καταδικάσω ε, απερίφραστα και να εκφράσω την ανησυχία μας τα όσα έγιναν στην Ονδούρα. Εγώ είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τη χώρα και την περιφέρεια τα τελευταία χρόνια ως αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας με την Κεντρική Αμερική και για μένα απολύτως σημαντικό την πρώτη μέρα τη συζήτηση πολιτική στο Κοινοβούλιο να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Δείχνουμε ότι του προσδίδουμε ε, θεμελιώδη σημασία. Είναι το πρώτο πραξικόπημα του 21ου αιώνα στην Κεντρική Αμερική και μεγάλο κρίμα. Επίσης, ε, θέλω να καταδικάσω, ε, καταδικάσω το πραξικόπημα, αλλά να πω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε το πραξικόπημα Τία αμυσελέτη να επανέλθει η συνταγματική τάξη στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προετοιμαστούν ε, με τρόπο σωστό και ε, νόμιμο οι εκλογές του Νοεμβρίου. Και τουλάχιστον προς στιγμή θα πρέπει να παγώσουν οι σχέσεις μας και οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Σε πάση περιπτώσει θέλω να ζητήσω όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοι και ε, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε έπραξαν να σταματήσει η βοήθεια στον εμπορικό τομέα εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια. Πέρα από όλα αυτά νομίζω θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σοβαρό το πραξικόπημα, ευθύνες έχουν πολλοί και σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι ε, δράστες από πίσω που δεν ξέρουμε τα ονόματά τους και αυτοργοί. Γι' αυτό θα πρέπει να στέλνουμε διεθνείς αντιπροσωπείες για να στηρίξουν τα κινήματα που αυτή τη στιγμή ξεκινούν στη χώρα για να μπορέσουν να ζητήσουν να επανέλθει η δημοκρατία που τους συναφέρεσαν τόσο ευεία. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα και κλείνει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων με τον κύριο Βίλι Μέγερ που θα μιλήσει εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις μέρες μετά το πραξικόπημο, η δική μου ομάδα αποφάσισε να στείλει εμένα στην Τεκουσιγκάλπα για να δω επιτόπου τις επιπτώσεις του στρατιωτικού αυτού πραξικοπήματος. Και είχα την ευκαιρία να δω με τα μάτια μου τα ίδια τι συνέπειε όπω όλα τα πραξικοπήματα. Δηλαδή, καταστολή, έλλειψη ελευθεριών. Συνάδελφοι βουλευτέ τη Βουλή που δεν ήταν υπέρ του ε, πραξικοπήματο έχουν συλληφθεί. Ε, είναι στη φυλακή ε, συνδικαλιστέ πολλοί τραυματίες ε, στα νοσοκομεία, απαγορεύση κυκλοφορίας κτλ. Εγώ χαίρομαι για την απάντηση του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η μόνη δυνατή απόκριση. Πρώτον, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι λένε οι οργάνωση των Αμερικανικών κρατών. Και πρέπει να σας πω ότι συναντήθηκα με το ε, γραμματέα του οργανισμού αυτού και είναι ξεκάθαρο στο μυαλό τους ότι ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση που είναι παράνομη του πραξικοπηματία Μιτσελέτη θα κηρυχθεί άκυρη. Δηλαδή, ο Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να στείλει παρατηρητέ σε εκλογέ που θα προκηρύξει αυτή η κυβέρνηση. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το κώδικα συμπεριφορά, αυτό το φύλλο πορεία τον μπούσουλα έτσι ώστε να μην ε, νομιμοποιήσει σε καμία περίπτωση την κυβέρνηση αυτή. Εμεί, λοιπόν υπό την έννοια αυτή δεν μπορούμε να στείλουμε παρατηρητέ που να τις ε, προκυρήσει τις εκλογές αυτή η πραξικοματική κυβέρνηση. Είναι αποφασιστική αυτή η εβδομάδα. Ο πρόεδρος Σελάγια που είναι ο μόνο πρόεδρο τη Οδούρα το ξεκαθάρισε. Έχει αφήσει διορία μία εβδομάδα και αν δεν λυθεί το θέμα αυτό μέσα στη εβδομάδα από διάλογο με την Κωνσταντίνα θα γυρίσει μόνο του. Λοιπόν, είναι ο μόνος νόμιμος πρόεδρος, αυτή είναι η απόφασή του και εγώ περιμένω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον συνοδεύσουν, να τον υποστηρίξουν, όπως το κάνει ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, τα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως οι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι, το τονίζω αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το ύφο. Απαιτητικό να επανέλθει η ε, ένομη τάξη, η συνταγματική τάξη, να γυρίσει ο πρόεδρος και αυτό να χαρακτηρίσει το κοινοβούλιο μας. Ελπίζω, συνάδελφοι, δε, να πάρουμε μια στεναρή απόφαση ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει κατηγορηματικά χωρίς κανένας είδους ε, απόχρωση ε, το πραξικόπημα και υποστηρίζουμε τους διεθνείς οργανισμούς στη δράση τους. Ευχαριστώ κύριε Μέγερ. Οι υπόλοιποι ομιλητέ τώρα που μιλούν προσωπικά για 1,5 λεπτό ο κύριος Καντέρ Αρίφ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να καταδικάσω, όπως και οι προλαλήσαντες, στεναρά το πραξικόπημα ε, κατά του Πρόεδρου Ζελαγιάς Αραράς, Συνδόρες. Παραβίαση του συνταγματικής τάξης που πρέπει να αποκατασταθεί. Στρατιωτική εξουσία που αυτό αυτοανήγγειλε αυτό ανήγγειλε νέο πρόεδρο είναι σκοτεινή περίοδος για την ιστορία της χώρας αυτής και προσβολή της δημοκρατίας απαράδεκτη. Χαιρόμεθα λοιπόν που αναβάλαμε, αναστήλαμε μάλλον τη συμμετοχή αυτής της χώρας στην, στον οργανισμό τη, χωρών Αμερικής, αλλά ανησυχώ κυρία Επίτροπε για τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με αυτή τη χώρα. Εδώ και πολλούς μήνες μία σύμβαση νέας γενναίας ε, τυχαίνει διαπραγμάτευσης. Το Χαιρόμαστε που οι διαπραγματεύσεις δεν έγιναν την περασμένη εβδομάδα και ακυρώθηκαν. Αλλά είπατε ότι θα αναστήλατε τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. Θα ήθελα να το ακούσω οριστικά από εσά, με βεβαιότητα δηλαδή. Και ε, ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό, Κομισιόν. Κυρία Επίτροπε, επίσης υπάρχει ένα θέμα, άλλο θέμα των γενικαβημένων προτιμήσεων. Πολλές ΜΚΟ έχουν μιλήσει για τις αυθαίρετες πράξεις βίας κατά και της λογοκρισίας από την εποχή του πραξικοπήματος. Οι μαρτυρίες είναι επαρκείς πρέπει να πω για να επιβεβαιώσουν ότι αυτό ο απαγγελθής πρόεδρος δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Μήπως θα μπορούσαμε να σταματήσουμε προσωρινά τις προτιμήσεις που έχουν χορηγηθεί στις Ονδούρες. Και δίνω τώρα το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Μελονσόν. Κύριε Πρόεδρε, οι ειρηνικές μας αρχές δεν πρέπει να μας οδηγούν να δίνουμε την εντύπωση ότι η συνταγματική κυβέρνηση και οι πραξικοπηματίες είναι ίδιοι στις Ονδούρες. Ζητούμε δηλαδή να είναι μετριοπαθείς και οι δύο πλευρές. Μα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην μεταχειριζόμαστε τις δύο πλευρές με τον ίδιο τρόπο. Οι μεν είναι εγκληματίες, πραξικοπαματίες. Θέλουμε να ζητήσουμε την αποκατάσταση και η επιστροφή του Ζελαγιά. Ε, όλη η Ήπειρος ουσιαστικά θέλει να τελειώσει με την περίοδο πραξικοπημάτων και δικτατοριών. Μετά την απόφαση του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανισμών πρέπει η Ευρώπη να αγωνιστεί και αυτή. Ε, ε, πρόκειται για αγώνα και όχι ρύθμιση. Είναι ιστορικός ο αγώνας. Θα πρέπει η Ένωση να διακόψει κάθε σχέση, εμπορική, πολιτική, κάθε διαπραγμάτευση με τους πραξικοματίες έως ότου ξαναβρει τη θέση του ο πρόεδρος Δελαγιάντη. Δεν υπάρχει τίποτα συμβιβαστικό που μπορεί να, να αποτελέσει λύση. Ακόμη και η Αμερική θα πρέπει να διακόψει τις σχέσεις της με αυτό το καθεστώς. Μόνο έτσι θα ανταποκραθούμε στις αρχές που επικαλούμε θα τόσο συχνά για να επικρίνουμε άλλους. Ευχαριστώ κύριε Μελανσόν. Και τώρα ακολουθούν Α, θέλω να πω ότι οι νέοι συνάδελφοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Είναι αυτό που λέγεται catch the eye. Δηλαδή, όποιον δύο πρόεδρο αυθόρμητα ζητάτε το λόγο, δύο συνάδελφοι, ξέρετε ότι έχετε ένα λεπτό έκαστο και θα σα κόψουμε το μικρόφωνο ακριβώ στα 60 δεύτερα. Πρώτο συνάδελφο που ζήτησε το λόγο, ο κύριο Σόνικ. Panie przewodniczący, sytuacja w Hondurasie wymaga kontynuowania przez Unię Europejską konkretnych i η κατάσταση στις Ονδούρες Χρειάζεται σταθερή δράση για να μπορέσει να επανέλθει το κράτος δικαίου στη χώρα και η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές να μην γίνει ακόμα πιο βίαιη. Γι' αυτό και υποστηρίζω την πρωτοβουλία του κυρίου Σαλαφράγκα να υπάρξει μια δυνατότητα να σταλεί μια αποστολή στις Ονδούρες στην Ονδούρα, συγγνώμη, ε, στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν καταφέρουμε να γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε ο πρόεδρος να μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά του και να εκτελέσει τη θητεία του μέχρι τέλους με κάποια αλλαγή στο Σύνταγμα ώστε να μπορεί και να επανακλήγει. Μια τέτοια λύση θα μπορούσε να δώσει κάποιες ελπίδες για σταθεροποίηση της κατάστασης και ίσως θα μπορούσε και να γίνει δεκτή. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι ως ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ως ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές προκειμένου να λιγοστέψουν οι μέρες του πραξικοπήματος στην ονδούρα και να επιστρέψει στη χώρα του ο πρόεδρος ελάγια να κλείσει επιτέλους ο κύκλος των στρατιωτικών πραξικοπημάτων στη λατινική και στην κεντρική αμερική. να αναλογιστούμε κύριοι συνάδελφοι τις μεγάλες προοδευτικές και δημοκρατικές αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από χώρες αλλαγές που ενισχύουν τις συνταγματικές και δημοκρατικές ελευθερίες που υπερασπίζονται την έννοια και την ουσία της πολιτικής έναντι της αχαλήνωτης τάσης της αγοράς να την εκτοπίσει που σπάνε τα μακρά δεσμά της νεοαπικιοκρατίας. γι' αυτό πιστεύω να αναλογιστούμε τις μεγάλες ευθύνες της ευρώπης για φιλειρηνική δράση στο διεθνές πεδίο και να αποκαταστήσουμε δεσμούς δημοκρατίας και αλληλεγγύης με τους λαούς και τις χώρες στην άλλη πλευρά του ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Λοιπόν, ολοκληρώνονται εδώ οι ομιλίες των βουλευτών για το θέμα αυτό και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπίλτ, εξ ονόματος του Συμβουλίου, για να απαντήσει. Μου είπαν ότι δεν θεωρεί σκόπιμο ούτε χρήσιμο να ξαναλάβει το λόγο η Επίτροπος, οπότε κύριε Μπίλτ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι όσοι μίλησαν, μίλησαν στεναρά για την προάσπιση του κράτους δικαίου και της συνταγματικής τάξης στη Λατινική Αμερική. Ό,τι και αν συμβαίνει δεν στέλνετε τους στρατιωτικούς για να ανατρέψουν τον συνταγματικά εκλεγμένο πρόεδρο. Άσχετα από την ιστορία και από το τι συμβαίνει. Όλοι είμαστε σαφέστατοι γι' αυτό. Αλλά για να επιληθεί η κατάσταση πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία, κάποιος συμβιβασμός. Και από ό,τι άκουσα από τον Σαραλαφράγκα και άλλους, όλοι θεωρούν ότι ο πρόεδρος Αρίες είναι κατά πάσα πιθανότητα ο καλύτερος άνθρωπος για να επιδιώξει αυτό το συμβιβασμό. Θα χρειαστεί χρόνο. Θα χρειαστεί χρόνο για να διαπραγματευτεί με εκπροσώπους και από τις δύο πλευρές αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να χαίρει τη υποστήριξή μα καθώς και της υποστήριξη των άλλων Αμερικανικών κρατών. Όσον αφορά τώρα τη φύση μιας λύσης, τα μέρη θα το συμφωνήσουν, αλλά από αυτό που είπα εξ αρχής, η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης είναι αυτό που αναζητούμε η επιστροφή του Προέδρου Σολάρ είναι απαραίτητη όταν μιλάμε για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Δεν θα φτάνει βέβαια, θα χρειαστούν και άλλα στοιχεία για να έχουμε αποκατάσταση συνταγματικής τάξης. Αυτό που ζητούμε λοιπόν είναι η επιστροφή του Προέδρου, η αποκατάσταση συνταγματικής τάξης, αλλά από μόνη της η επιστροφή του Προέδρου δεν θα επαρκεί. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ σημαντικά για τις σχέσεις μας με αυτή τη χώρα, για την ανάπτυξη αυτής της χώρας και για την αξιοπιστία της δημοκρατίας σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Μετά την ομιλία του Προεδρεύων Συμβουλίου ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή και σε ό,τι αφορά την ε, Ανακοίνωση των προτάσεων διάσκεψη του Προέδρου για του ορισμού στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Πρέπει να σα πληροφορήσω ότι θα σας διαβιβαστούν όλα αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο ίδιος κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης και επίσης πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεση ε, ε, τυχών τροπολογιών ολοκληρώνεται απόψε στι 7.